I uh, Ας αρχίσουμε παρακαλώ. Ας αρχίσουμε με τις αποφάσεις που πήραν χτες οι συγητές ή μάλλον διορθώνει πρόεδρος οι σύντονιστές. Σχετικά με γνωμοδοτήσεις, ή νομοθετικές γνωμοδοτήσεις πρώτα απ' όλα. Δύο γνωμοδοτήσεις έχουμε για την αλλαγή στο καθεστώς του Μαγιότ. Το πρώτο είναι η προστασία των ζώων, η υγιεινή, η λύση κτλ. Το δεύτερο είναι η δημόσια υγεία. Και οι δύο αυτές γνωμοδοτήσεις πάνε στους σοσιαλιστές. Στη συνέχεια έχουμε τις ε, αποφάσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία που πάνε στο ΕΛΚ. Κάθε φορά έχουμε και το Ταμείο Προσαρμογής, αλλά δεν έχουμε χρόνο για να κάνουμε αυτό που κάνουμε συνήθως, που είναι η επιστολή του, της Πρόεδρου για να μην καθυστερήσει όλη η διαδικασία. Υπάρχει πάντως η δυνατότητα οι συντονιστές να το αναλάβουν. Στη συνέχεια έχουμε τη γνωμοδότηση στην Πράσινη Βίβλο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Οικονομία, ΕΛΚ. Έχουμε μετά την γνωμοδότηση ίδιας πρωτοβουλίας πώς η Ευρώπη μπορεί να συνεισφέρει σε ένα καλό κλίμα για τις επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις startup προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, των αναλαμβάνουν οι σοσιαλδημοκράτες. Επίσης, σε πρόγραμμα δράσης για την αηφόρο ανάπτυξη Άλντε και συζητήσαμε και κάτι ακόμα. Πώς φέτος θα ασχοληθούμε στην Επιτροπή μας για τις δημοσιονομικές τροπολογίες και για το 2013 και τη γνωμοδότηση για τον προπολογισμό το 2014. Συμφωνήσαμε λοιπόν την εξής διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια κάνουμε το ίδιο εξάλλου. Αποφασίσαμε λοιπόν να δώσουμε εντολή στον εισηγητή και την πρόεδρο να ξεκινήσουν με μια βάση υπόθεσης ότι θα αποδεχτούμε τον προπολογισμό σαν το ελάχιστο που μπορεί να χρειάζεται η Ευρώπη. Και εφόσον υπάρξουν περικοπές, όπως συμβαίνει συνήθως από το Συμβούλιο, το ο Πρόεδρος και συγητής θα προσπαθήσουν να επιστρέψει στην αρχική του μορφή ο προπολογισμό. Είναι αυτό που κάνουμε τα τελευταία χρόνια έτσι κι Πρόεδρος και εισηγητή. Συμφωνήσαμε επίσης και δεχτήκαμε το αίτημα του Derek Βόν σε σχέση με την έκθεσή του. Ζήτησε ένα σημείωμα ενημέρωσης από το Τμήμα Πολιτικής και για τις εξωτερικές μελέτες θα αποφασίσουμε το Σεπτέμβριο. Οι συντονιστές θα σκεφτούν κατά τη διάρκεια του θέρους σε σχέση με τις μελέτες αυτές. Έχουμε και ένα αίτημα από το ΕΛΚ να ακυρώσουμε τον Οκτώβριο την αντιπροσωπή μας που θα πήγαινε στη Βουλγαρία, κάτι το οποίο έγινε αποδεκτό και συμφωνήσαμε ότι θα επανέλθουμε το Σεπτέμβριο. Ακούστηκαν διάφορες προτάσεις αλλά δεν πήραμε καμία απόφαση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την Βουλγαρία και μετά που θα πάμε, αν θα πάμε κάπου, στο διάστημα αυτό που προβλεπόταν αρχικά η επίσκεψη στη Βουλγαρία. Και τώρα πάμε στο σημείο 18 στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε μαζί μας τον Ραφαέλ Γκουλέ που είναι ε, επικεφαλής της ε, μονάδας ε, που είναι υπεύθυνη για την Αυστρία, τη Σλοβενία και την Κροατία. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στο Ραφαέλ Γκουλέτ προκειμένου να μας ενημερώσει τι κάνει η Κροατία σε σχέση με το Ταμείο Συνοχής, τα κονδύλια συνοχής και τι προκλήσεις αντιμετωπίζουμε τώρα τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η Κροατία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε την ευκαιρία να εξηγήσουμε το τι γίνεται σε σχέση με την προετοιμασία της πολιτικής συνοχής ε, στην Κροατία ε, κάτι το οποίο είναι βεβαίως πολύ περίπλοκο γιατί μιλάμε για τρεις διαφορετικές περιόδους ε, που θα περάσουν πάρα πολύ γρήγορα. Μέχρι 1η Ιουλίου υπήρχε προενταξιακή βοήθεια ακριβώς για να προετοιμαστεί για την διαρθρωτική πολιτική και τώρα είναι από 1η Ιουλίου στο νέο καθεστώς πολιτικής συνοχής και μπορούμε να πούμε και πρέπει να αναγνωρίσουμε πως οι προσπάθεια της τον τελευταίο μήνα ήταν ακριβώς για να προετοιμαστεί αυτή η μετάβαση. Να ξεκινήσω λοιπόν με το μέσο αυτό της Ανατολικής Γειτονίας. Είχαμε τρία προγράμματα, ένα για μεταφορές, ένα για περιβαλλον και ένα για περιφερειακή ανταγωνιστικότητα το οποίο βέβαιω είναι αυτό το οποίο κάναμε και με άλλες ε, χώρες ε, προένταξης και βεβαίως ε, τα προγράμματα αυτά περιέχουν ένα σημαντικό στοιχείο στο οποίο μαθαίνει κανείς κάνοντας και μπορούμε να πούμε πως είναι ακριβώς το μέσο ανατολικής συνοχής πιο, πιο συγχωρείτε, πιο προσαρμοσμένο σε ζητήματα όπως ο πολιετής ε, προγραμματισμός ε, και ο προγραμματισμός με βάση κάποια διάρθρωση. Λοιπόν, το ποστό απορρόφησης τα τελευταία χρόνια ήταν 40% αλλά αν βγάλουμε τις προκαταβολές ήταν 26% μόνο, κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί και ικανοποιητικό δεδομένο του ότι η εφαρμογή ξεκίνησε μόλις το τέλος του 2008. Γιατί αργήσαμε τόσο, γιατί χρειαζόταν χρόνος για να υπάρξει κάποια προετοιμασία των δομών διαχείρισης και ακόμα και η εφαρμογή η πραγματική των έργων ξεκίνησε τέλος 2009, αρχές 2010 και έχουμε εδώ πέρα και κάποια αντίγραφα του περιοδικού μας, βεβαίως, όπου καλωσορίζουμε την Κροατία, αλλά φαίνονται και κάποια έργα που συγχρηματοδοτούμε. Παραδείγματο χάρη, θα θέλαμε να δώσουμε ένα παράδειγμα, για το κέντρο εμπορευματοποίησης ε, των βιολογικών ε, επιστημών ε, σε ένα πανεπιστήμιο της Κροατίας. Οπότε στο τέλος της ε, προγραμματικής ε, περίοδου συμφωνήσαμε τα επίσημα προγράμματα συνοχής 2007-2013 ε, να βασιστούν στην εμπειρία που είχαμε στην Ανατολική Γειτονία γιατί, γιατί λίγο πολύ θα ισχύσουν τα ίδια συστήματα διαχείρισης και ελέγχου κάτι το οποίο σημαίνει πως όλα τα Υπουργεία θα παραμείνουν υπεύθυνα για τα προγράμματά τους π.χ το Υπουργείο Μεταφορών για τα ζητήματα μεταφορών και ναυτιλίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος αντιστοίχω για το περιβάλλον. Το μόνο ζήτημα ήταν η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα που πήγε από το Υπουργείο Οικονομίας στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τι γίνεται λοιπόν. Τα προγράμματα αυτά επεκτείνονται ουσιαστικά μέχρι το τέλος τη προγραμματικής ε, περίοδου συν άλλο ένα έτος μέχρι το 2016 για να υπάρχει περισσότερος χρόνος ε, για την εφαρμογή και βεβαίως με τις ίδιες προτεραιότητες αλλά με ενοποιημένους δείκτες και παραπάνω κονδύλια. Οπότε να σας πενθυμίσω πως ε, μιλούσαμε για 538 εκατομμύρια ευρώ από την Ανατολική Γειτονία, στα οποία θα προσθεθούν 450 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Πώς θα μοιράζουμε το πρώτο πρόγραμμα της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας είναι καθαρά ΕΤΠΑ ε, και υποστηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κοινοτομία και ανάπτυξη κτλ. Το πρόγραμμα των μεταφορών επίσης τελείως ΕΤΠΑ και συγχρηματοδοτεί μόνο σιδηρόδρομους, ε, πλωτούς ποταμούς κτλ. Το περιβάλλον είναι μόνο στο Ταμείο Συνοχής για κυρίως ζητήματα βιολογικού καθαρισμού και κοινωνικής ένταξης κλπ. Και βεβαίως υπάρχει, υπάρχουν και κάποια προγράμματα διασυνοριακά με την Ουγγαρία και τη Σλοβενία και άλλα περιφερειακά προγράμματα. Οπότε ποια είναι τα επόμενα βήματα για το 2007-2013. Έχουμε συνεργαστεί στενά με τους Κροάτες και αναμένουμε βεβαίως την επόμενη έκδοση του, των εθνικών αρχών και βεβαίως θα πρέπει να δούμε και τον Ιούλιο τις ε, αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν και ελπίζω να υιοθετηθούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού από την Κομισιόν και βεβαίως ε, θα πρέπει να έχουμε και έτοιμα τα συστήματα διαχείρισης ε, και ελέγχου και ελπίζουμε η Κομισιόν να μπορέσει να το διευθύνσει πριν από το τέλος του έτους. Οπότε, δεν ναι, ήταν κακή αρχή, αλλά οι προκλήσεις είναι τεράστιες και θα απαιτήσουν πραγματικά κάποιες θεσμικές προσαρμογές στην Κροατία. Όπως είπα λοιπόν η Κροατία εντάσσεται στο τέλος αυτής της ε, προγραμματικής περίοδου και είναι δύσκολο για την κροατική διοίκηση να προετοιμαστεί και για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης δηλαδή από το 2014 με 20. Βεβαίω τώρα διπλασιάζονται τα κονδύλια, το εξάμεινο που απομένει μέχρι το τέλος του έτους, αλλά αν δείτε ολόκληρη την περίοδο 2007-2013, θα έχουμε έναν ε, οκταπλασιασμό. Ουσιαστικά μιλάμε για 8 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή συνολικά ΕΤΠΑ και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και άλλα 2 δισεκατομμύρια από το Γεωργικό Ταμείο και 200 εκατομμύρια από το Ταμείο της Αλίας. Υπάρχει λοιπόν αρκετά μεγάλη επιτυχία των κρατικών αρχών και προσπαθούμε να συνεργαστούμε για να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα. Βεβαίως ε, το πρώτο δεν θα σας προξενήσει εντύπωση αφορά την διοικητική ικανότητα των Υπουργείων η οποία έχει βελτιωθεί αλλά Οπωσδήποτε δεν ε, έχουμε φτάσει στο τέλος διαδικασίας. Ελήφθη απόφαση να προσληφθούν γύρω στους ε, πάνω από 200 διαχειριστές των ταμείων πέρσι οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί ακόμα βεβαίω για λόγους προϋπολογισμού Ο άλλος παράγον που θα ήθελα να αναφέρω είναι η συντονισμένη διυπουργική συνεργασία ε, που είναι μια πρόκληση για την ε, Κροατία και αυτό το βλέπουμε και για τις μελλοντικέ περιόδους καθώς θα πρέπει να δοθούν οι σωστές ε, προτεραιότητες. Το τρίτο στοιχείο είναι απλοποίηση των διαδικασιών Βλέπουμε έτσι μετάβαση από κάποιους κανόνες σε κάποιους άλλους, αλλά υπάρχει κάποια τάση μετά ανατροπή των αποφάσεων, κάτι το οποίο δεν κάνει τόσο εύκολες τις, ε, τη λειτουργία της ε, διοίκησης στην Κροατία. Βεβαίω όλα αυτά είναι καινούργια στη διοικητική λειτουργία της χώρας, αλλά αυτό έχει γίνει και άλλο στο παρελθόν. Και έχουμε κάποια επιτυχία. Π.χ. 6 Ιουνίου υπήρχε μια διάσκεψη των εταίρων στο Ζάγκρεπ για το μέλλον, αλλά οπωσδήποτε μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα και βεβαίω το ζήτημα είναι να υπάρχει ειδοποίηση για μεγάλα έργα και βεβαίω η αύξηση των δυνατοτήτων στο τοπικό επίπεδο και στο επίπεδο του Υπουργείου και χαιρόμαστε για το ότι η Κροατία εδώ και ένα χρόνο χρησιμοποιεί τη στήριξη του Τζάσπερς οπότε όλα τα μεγάλα έργα που έχουν υιοθετηθεί μέχρι στιγμής έχουν ωφεληθεί και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Ε, τέλος ε, να πω λίγα λόγια για την προετοιμασία της περίοδου 2014-2020. Ξέρω πως έχουν λάβει χώρα όλες οι σημαντικές ε, ψηφοφορίες. Τεράστια πρόκληση, ούτως ή άλλως 8 δισεκατομμύρια, τεράστια πρόκληση για τη διοίκηση. Όπως και με τις άλλες χώρες ζητήσαμε από την Κομισιόν ένα έγγραφο θέσεων και οι τέσσερις προτεραιότητες που ζητάμε από την Κροατία είναι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σύμφωνα με το πρόγραμμα 2020. Το δεύτερο είναι η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Ε, αύξηση των δεξιοτήτων μείωση της φτώχειας, ε, τρίτη προτεραιότητα είναι προστασία του περιβάλλοντος ε, και τέλος ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας. Είναι νωρίς ακόμα για να γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι επιλογές. Είναι προφανές πως με την Κροατία έχουμε προχωρήσει αρκετά στην διαδικασία, αλλά ότι αντιλαμβανόμαστε θα υπάρχουν τρεις διαχειριστικές αρχές ε, Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εργασίας ε, και Απασχόλησης οπότε θα έχουν μια κεντρική προσέγγιση για ολόκληρη τη χώρα Νομίζω φτάνουν αυτά για την ώρα και είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ πολύ το Γιάνν Όλμπριχτ πρώτα. Όποιος θέλει το λόγο, παρακαλώ. Μετά. Ναι, έχω μία ερώτηση. Γιατί έχω χαθεί λιγάκι με τους νέους διακανονισμούς. Γιατί είχαμε μια δύσκολη συζήτηση για τα 400 εκατομμύρια για την Κροατία που λείπανε. Και έπρεπε να γίνει. Τώρα που είμαστε στα τέλη της περίοδου 2013, από ό,τι έχω καταλάβει, στο τέλος θα έχουμε τα νέα λειτουργικά προγράμματα βάσει του κανονισμού 17-13 με 8 εκατομμύρια. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, προς όφελος των ε, κρατών φίλων ρωτάω δηλαδή, αυτά τα 8 εκατομμύρια πού είναι, από πού θα έρθουν γιατί έχουμε πρόβλημα με τον προπολογισμό του 2014. Έχουμε έλλειμμα για το 2013. Οπότε, έρχομαι στη δεύτερη, θα ισχύσει ο κανόνας του νησιν 3 για την Κροατία. Νησιν 3 δεν θα είναι, ή θα είναι νησιν 2 ή νησιν 2,5. Νομικά μιλώντας δηλαδή, τι θα ισχύσει. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Μπορεί να υπάρχει βέβαια κάποια μετάβαση, κάποιος μηχανισμός μετάβασης. Αλλά το λέω για όλους μας και κυρίως για τους Κροάτες φίλους. Πώς οργανώνονται όλα αυτά, γιατί το 2014, 2015 και 2016 θα πρέπει να γίνουν πληρωμές. Ελπίζουμε να έχουμε την ευελιξία. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε περισσότερα πράγματα για το πώς θα οργανωθούν όλα αυτά. Ευχαριστώ. Και από την Κροατία έχουμε τη συνάδελφο. Για πείτε μας ε, ποια είσαστε, να σας γνωρίσουμε. Είμαι η Βάνα Μάλετζιξ και όντως είμαι νέα ευρωβουλευτής από την Κροατία. Σας ευχαριστώ όλους για τον τρόπο που μας υποδεχτήκατε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετείχα σε όλες αυτές τις διαδικασίες στην Κροατία για τον διακανονισμό του ΙΠΑ και τις προπαρασκευαστικές δράσεις όσον αφορά τη συνοχή. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω στην ερώτηση του Γιάνν, φαντάζομαι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το κάνει. Θα ήθελα όμως εγώ να ρωτήσω δύο άλλα πράγματα. Πρώτον, σε σχέση με την δυνατότητα να πάρει προκαταβολές η Κροατία για αυτή την περίοδο για την Κροατία. Είναι πολύ σημαντικό μέχρι τα τέλη του 2013 να πάρει αυτά τα χρήματα για να υπάρχει ρευστότητα. Και θέλω επίσης να ξέρω Φαντάζομαι τον Ιούλιο θα πάρετε την περιγραφή της διαχείρισης. Μετά θα σας πάρει χρόνο να το μελετήσετε και να δείτε αν θα δώσετε την άδεια για να αρχίσει η εφαρμογή, όχι. Και κάτι άλλο όσον αφορά τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την περίοδο 2014-20. Όλοι είμαστε επικεντρωμένοι στο δεύτερο εξάμεινο του 2013. Και φυσικά και είναι πολύ σημαντικό αλλά δεν έχω καταλάβει, υπογραμμίσατε βέβαια εσείς ότι αυτή η διαδικασία ε, συνεργασίας και εταιρική σχέσης πρέπει να ενισχυθεί, όμως σε σχέση με την Κροατία αυτό δεν το βλέπω. Και για τις διοικητικές ικανότητες προχωράμε σε στρατηγικές και προγράμματα δράσης για την οργάνωση στρατηγικών ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά για την χρηστή οικονομική διαχείριση και την εφαρμογή παρετέρω. Ο Βίκτορ Ποστινάρο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θυμάμαι το 2008, άνοιξη του 2008, μόλις είχα εκλεγεί ευρωβουλευτής στη Ρουμανία. Συναντήθηκα λοιπόν με αξιωματούχους και δημοσιογράφους από την Κροατία, οι οποίοι με ρώτησαν για τη δικιά μας εμπειρία που τη θεώρησαν ε, ε, καλή. Όχι βέβαια για να μεταφέρουμε την ε, δικιά μας εμπειρία σε αυτούς, γιατί τότε θα έλεγα ότι δεν πήγαιναν πολύ καλά τα πράγματα, αλλά αν μη τι άλλο έδειξαν ότι θέλαν να λάβουν υπόψη τους όλες τις εμπειρίες και να καταλήξουν σε συμπεράσματα για το τι τελικά θα ταιριάσει καλύτερα στις ανάγκες της Κροατίας. Χωρίς λοιπόν να γνωρίζω περισσότερο τις εξελίξεις στην Κροατία, θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, πώς αξιολογείται σήμερα τη θεσμική και διοικητική ικανότητα της χώρας να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις εφαρμογής της νέας πολιτικής συνοχής. Γιατί αν δούμε τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την εμπειρία της Πολωνίας και άλλων για διοικητική και θεσμική ικανότητα, έχει αποδειχτεί ότι αυτή είναι ζωτική σημασία. Πώς έχει λοιπόν αυτό στην Κροατία. Δεύτερον, η Κομισιόν πώς θα φροντίσει για την επόμενη περίοδο. Δεν θα υπάρξει αστάθεια στην Κροατία ούτε πολιτική ανάμειξη στον τομέα των εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Γιατί και πάλι από την εμπειρία που έχω από τη δικιά μου χώρα, κακή εμπειρία στη Ρουμανία, η αστάθεια των θεσμών δημιουργεί τεράστια προβλήματα όπως επίσης και η πολιτική ανάμειξη στον τομέα των εμπειρογνωμόνων. Καταστροφικές είναι οι συνέπειες. Θέλω λοιπόν να ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν μη τι άλλο, έχει υπόψη τις, τις καλές και τις κακές πρακτικές, έτσι ώστε τώρα η Κροατία ή άλλες υποψήφιες χώρες στο μέλλον θα μπορούν να έχουν ισχυρούς και αξιόπιστους θεσμούς και διοικητικές ικανότητες. Με πυρογνώμονες η Κροατία μπορεί να τα καταφέρει πολύ καλύτερα μια που γνωρίζει και τη συμπεριφορά της δημόσιας διοίκησης, την οτροπία, τις αντιδράσεις του κόσμου. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην Κροατία και να ξέρετε ότι χρειαζόμαστε πολλά καλά παραδείγματα για τα Δυτικά Βαλκάνια για να δείξουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Το λέω με κάθε σεβασμό πρέπει οι άλλες υποψήφιες χώρες να πάρουν παράδειγμα, να δούνε δηλαδή ένα καλό παράδειγμα για να ετοιμαστούν και αυτοί θεσμικά και διοικητικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Βίκτορ. Ο Γιάννης Νίλσον έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα καλώς ήρθατε και εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βλέπω ότι η Κροατία αποτελείται από 21 διοικητικέ αρχές. Η διαχείριση των διορθωτικών κονδυλίων όμως θα γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι αποφάσεις για τα προγράμματα θα λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Μαρίτερες Σάντσε Σμιθ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, συνάδελφε, από την Κροατία. Βρισκόμαστε σε μια επιτροπή που είναι ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον της Κροατίας. Ήθελα να μιλήσω λίγο για την ανταφική συνεργασία, διότι κατανοούμε ότι μέχρι τώρα ακούσαμε για την ικανότητα της χώρας να αξιοποιήσει αυτά που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ε, τομέα των ε, περιφερειακών ταμείων και των διαφορετικών ταμείων και πιστεύω ότι η εδαφική συνεργασία θα λαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία είτε είναι διασυνοριακή, είτε διαπεριφερειακή, είτε σε ό,τι αφορά το διαπεριφερειακό στοιχείο, τι προσέγγιση ακολουθήσατε. Διότι για μια χώρα που προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και θετικών εμπειριών λαμβάνει μεγάλη σημασία. Με χώρες όπως η Ρουμανία, που ήταν οι τελευταίες που προσχώρησαν, από τις τελευταίες που προσχώρησαν, σίγουρα μπόρεσε να αποφεληθεί από τις προηγούμενες εμπειρίες των άλλων κρατών. Τι διδάγματα λοιπόν αντλήσατε από το παρελθόν και στα κονδύλια. Στα κονδύλια που σας αποδόθηκαν είδαμε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ να προέρχονται από τα διευθυντικά ταμεία. Ε, αξιοποιήθηκαν αυτά πλήρως, δαπανήθηκαν και αν όχι γιατί. Ευχαριστούμε Μαριτερέ, ο, ο κ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω μια πολύ απλή ερώτηση που έχει να κάνει με την αρχή της εταιρική σχέσης. Το ανέφερε ευθύ εξ αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό είναι μεγάλη πρόκληση για την τρέχουσα περίοδο. Ήθελα λοιπόν η Επιτροπή ή τα μέλη από την Κροατία να μου πούν Τι έγινε ως τώρα με τα, προγράμματα, με τα λειτουργικά προγράμματα και με τη συμμετοχή των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Πώς συμμετείχαν στο σκέλος της ε, πολιτικής συνοχής. Πρόεδρος, δεν έχω κάποιον άλλο στον κατάλογο των ηγορτών. Ραφαέλ, εάν θέλεις, γιατί και για να περιμένεις και τη συνάδελφα από την Κροατία, γιατί καταλαβαίνω ότι και εσύ χαίρεσαι που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Εάν θέλεις λοιπόν να ακούσουμε μετά από σένα την συνάδελφα από την Κροατία. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για τον προπολογισμό, ίσως δεν ήμουν σαφής. Τα 8 δις ήταν το κονδύλι για το 14-20, για αυτό το διάστημα. Αυτό ήταν μέρος της συμφωνίας του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τον κανόνα MP3 Ήδη στη Συμφωνία Εταιρική Σχέση είχαμε τον κανόνα αυτό και η συνθήκη προσχώρηση θα επιτρέψει τεχνικώ αυτό το νέο εξάμενο να παρατείνει την ισχύ του κανόνα. Δηλαδή η Κροατία για έναν ακόμη χρόνο μέχρι το τέλο του 2016 μπορεί να αποφεληθεί από αυτόν τον κανόνα. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση που έγινε για το σύστημα διαχείρισης ναι, και φέτος θα μα αποσχολήσει αυτό και θα κοιτάξουμε να υπάρξει συμμόρφωση με του κανονέ μέχρι το τέλος της χρονιάς για να μπορεί να παίρνει ακόμα χρηματοδότηση η Κροατία. Αυτά ίσχυαν μέσα του διαστηματο 2007 2007-2013, οπότε και τώρα τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου παρατείνονται. Γι' αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερω η απόφαση τη Κροατία. να βασιστεί στα προγράμματα και στο διάστημα 2007-2013 για το επόμενο το 2014-2020 αξιοποιώντα τις υποδομές του, της τη e της Συμφωνίας Τρικής Σχέσης αλλά συζητήσαμε και με τις διοικητικές αρχές της Κροατίας, με τις ελεγκτικές αρχές και τις δικές μας υπηρεσίες και ελπίζουμε ότι αυτό το οποίο θα έχουμε τον Ιούλιο θα είναι καλής ποιότητας. Πριν όμως το δω δεν μπορώ να προδικάσω το αποτέλεσμα. Πρέπει να το έχει αποτιμήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την ε, συμμόρφωση. πριν ε, αποφανθούμε και θέλουμε να αποφύγουμε προβλήματα ρευστότητα για την Κροατία τον πρώτο χρόνο τη προσχώρηση. Όσο για το διάστημα 14-20, αυτό ήταν ένα από τα ε, ένα στοιχείο τη ανάλυση μα όταν αξιολογούσαμε τα προηγούμενα προγράμματα, διότι δεν είχαν ακόμα αρκετέ δυνατότητε στα Υπουργεία. Τώρα όμως έχει δοθεί έμφαση στην προετοιμασία για το διάστημα 14-20. Και φαίνεται να μπορούμε να γυρίσουμε τη σελίδα αυτή της ιστορίας. Είμαστε λοιπόν βέβαιοι ότι οι κροατικές αρχές, σε αντίθεση με το παρελθόν, θα δώσουν μεγάλη έμφαση στο να προετοιμαστούν σωστά για το 2020 και στα έγγραφα που απεικονίζουν τις ε, διάφορες, την κατάσταση στις, στις διοικητικές αρχές, αυτά που παρουσιάσαμε τον Γενάρη, είναι σαφές ότι ήδη υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για τις στρατηγικές επιλογές και έχουμε και μια συνάντηση με προσώπους της Κροατίας την ερχόμενη Τρίτη. Οπότε θα διαμορφωθεί τελικά η στρατηγική αυτή. Φυσικά λείπει ακόμη και το έγγραφο αυτό είναι μια πρώτη επικόνηση του τι περιμένουμε, αλλά δεν αρκεί. Θα πρέπει και το Τζάσπερ που βοήθησε ως τώρα τους Κροάτες να καταρτήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική για τις μεταφορές, να αξιοποιηθεί. Θέλουμε η στρατηγική να είναι έτοιμη για του χρόνου. ή για τα ευθύ δίκτυα και τη στοιχειατική στρατηγική. Και στο περιβάλλον πρέπει να γίνουν μεγαλύτερε προσπάθειε. Στι διοικητικέ ε, δυνατότητε έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που βρίσκουμε πολύ θετικό είναι ότι στι πρώτε συζητήσει με την Κροατία για την προετοιμασία 2014-2020 είπαν ότι και κατάλαβαν ότι θέλουμε να πάρουν πολύ σοβαρά το στόχο που είχε τεθεί για το 2011 για τι διοικητικέ δυνατότητε και τι συνήθει δυνατότητε. Εδώ θέλουμε πραγματικά να τους ενισχύσουμε, οπότε πρέπει να δοθεί σωστή εστίαση στο θέμα. Η Κροατία προσπαθεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. ακούει πολλές διαφορετικές απόψεις από πολλές πηγές και στηρίζονται και πολλές εταιρείε, όπως είχαν στηριχθεί ως τώρα από την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και από τη Λιθουανία και από την Ουγγαρία ε, λαμβάνει στήριξη και από αλλού, αλλά φοβούμαστε ότι εάν δεν έχουν απαρκή στήριξη τα Υπουργεία δεν θα λειτουργήσουν απαρκώς. Ακόμη και αν το προϊόν, το αποτέλεσμα από άλλα κράτη-μέλη είναι καλό, δεν μπορεί να αξιοποιήσει πλήρω. Δεν υπάρχει λοιπόν επαρκή πρόοδο για την ε, πλήρη βελτίωση των δυνατοτήτων στα ίδια τα Υπουργεία. Σε ό,τι αφορά την αστάθεια, ω τώρα, ναι, υπάρχει ο κίνδυνος ελοχεύει, αλλά το περιβάλλον έχει σταθεροποιηθεί μάλλον. Ελπίζω ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί, αλλά έχετε δίκιο. Θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ζήτημα. Για τις περιφέρειες για το πώς αυτά γίνονται αντικείμενα διαχείριση σε εθνικό επίπεδο. Ναι, λόγω της έλλειψης διοικητικών δυνατοτήτων είναι δύσκολη η κεντρική διαχείριση από την πλευρά των Υπουργείων. Όμως, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι οι 21 κομιτείες κάνουν ό,τι μπορούν ε, καλύτερο για να ετοιμάσουν τα προγράμματα και για τη συμμετοχή των αρχών, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Δύο στοιχεία εδώ. Υπάρχουν εκπρόσωποι των συλλόγων τοπικής αυτοδιοίκησης σε κάθε ε, επιτροπή ελέγχου, παρακολούθησης μάλλον, οπότε είναι μέρος της διαδικασίας υλοποίησης, συμμετέχουν πλήρως. Και στις 6 και 7 Ιουνίου υπήρξε μια μεγάλη συνδιάσκεψη για την προετοιμασία για το 2020 με συμμετοχή των αρχών τοπική αυτοδιοίκηση και των εκπροσώπων των διαφορών κομιτεών. Δεν λέω ότι αυτό αρκεί, αλλά οι διοικητικέ αρχέ κατάλαβαν το πλεονέκτημα του να είναι ανοιχτέ σε νέε ιδέε και να εφαρμόζουν νέε λύσει. Και μια τελευταία παρατήρηση. Αυτό που είπε η κυρία Σάντσε Σμιθ για την ε, διαπεριφερειακή συνεργασία. Η Κροατία το γνωρίζει αυτό και είναι και αρκετά ενεργή, όπω με τη στρατηγική του Δούναβη. Προσπάθησε να υποφεληθεί από εμπειρίες και θετικά διδάγματα από άλλους και ασχολείται και με τις προηγούμενες στατικικές για την Αδριατική λόγου χάρη, την ε, στατική της Ένωσης για την Αδριατική. Είναι σημαντικό να υποφελείται κανείς από τις εμπειρίες άλλων. Επειδή λοιπόν ασχολήθηκα με την Κροατία, αλλά άλλοτε και με τη Σλοβενία και την Αυστρία, το Φεβρουάριο συνοργανώσαμε μία σύνοδο για τη στρατηγική του Δούναβη και είναι σίγουρα ένα πρώτο βήμα. Δεν αρκεί, δεν είναι το μόνο, αλλά όντω θέλουμε οι συνεργάτε μα, οι εταίροι μα να, να υποβοηθούνται για να βρουν την κατάλληλη κατεύθυνση. Και τον ε, περασμένο Δεκέμβριο είχαμε ένα σεμινάριο για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων για τις δημόσιες προμήθειες. Ήταν ένα πρώτο στάδιο, δεν λέω ότι αρκεί, αλλά ήταν μια πρώτη φάση στην όλη διαδικασία. Κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο και για του υπόλοιπου, δηλαδή, από τι θετικέ εμπειρίε των προηγούμενων. Ευχαριστώ. Ε, Ιβάνα, θέλει και εσύ να σχολιάσεις. Σα ευχαριστώ. Να πω ότι είμαι ευγνώμων που προβλέψατε αυτή τη συζήτηση στην ημερήσια διάταξη για το πώς έχουν τα πράγματα στην Κροατία και νομίζω ότι θα πρέπει και σε επίπεδο κοινοβουλίου να ενημερώσουμε. Οπότε βάσει τη συζήτηση αυτή θα κάνω ό,τι μπορώ για να προτείνω τέτοιου συζητήσει στο Κροατικό Κοινοβούλιο. Από πολιτική άποψη είναι σημαντικό να έχουμε σωστή υλοποίηση τη πολιτική συνοχή. Για την Κροατία η πολιτική συνοχή έχει τεράστια σημασία. Βαρύνει ιδιαίτερα στη χώρα λόγω των κονδυλίων που επενδύονται αλλά και ως προς τις προτεραιότητες και την στρατηγική, το στρατηγικό σχεδιασμό. Κάτι που θα πρέπει πλέον να αποσχολήσει όλη τη χώρα. Σίγουρα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η μορφή διαλόγου μεταξύ κεντρικής και περιφερειακών κυβερνήσεων. Όλοι καταλαβαίνουν αυτή την ανάγκη διότι υπάρχουν μεν εθνικά προγράμματα, αλλά είναι πολύ δραστηρίε και οι περιφέρειε, οι κομιτείε μα και θέλουν να συμμετέχουν, θέλουν να είναι μέρο τη διαδικασία. Καθημερινά στην Κροατία ε, θέτουν ερωτήσεις, ερωτήματα. Ζητούν πληροφορίε για τα λειτουργικά προγράμματα, για τι στρατηγικέ και ούτω καθεξή. Αυτό που πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο είναι πρώτα απ' όλα να κάνουμε κάποιε στρατηγικέ επιλογέ. Διότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά τι θεματικέ προτεραιότητε του 2013-2020 2011-2013, πολλές είναι ιδιαίτερα ελκυστικέ και κάθε νέο μέλος δεν είναι αναγκαστικά σε θέση να διαλέξει σωστά. Ε, κάποιοι πέφτουν στην παγίδα, στο κοινοβούλιο λόγω χάρη, να διαλέξουν όσο περισσότερα γίνεται και δεν επικεντρώνονται στη σωστή ανάπτυξη. Οπότε ελπίζω ότι με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτή τη διαδικασία η Κροατία θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Επίσης βλέποντας το ύψος των κονδυλίων για την περίοδο 2014-2020 προβλέπονται για μας 8 δις από την πολιτική συνοχή. Αλλά υπάρχουν και γεωργικά κονδύλια για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η ανάπτυξη της υπαίθρου προσωμιάζει με την ε, συνοχή, με την πολιτική συνοχή. Σε μια επταετία λοιπόν έχουμε ένα πολύ σημαντικό μέρος του κρατικού προπολογισμού και αυτό είναι μεγάλη σημασία και για την οικονομική αύξηση και την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Είναι σημαντικό όλα αυτά να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και να επιταχύνουμε και εμείς την ανταξιακή μας ε, προσπάθεια. Κάτι που φαντάζομαι ότι είναι κοινό σκοπός ε, και των υπόλοιπων κατομελών και της Κροατίας. Για την ώρα δεν συμμετέχουμε στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, αλλά θα πρέπει κάπως να συνεισφέρουμε αφού επιτύχουμε μερικά αποτελέσματα. Αφού δηλαδή έχουμε οριμάσει αρκετά ώστε να μπορούμε να συμμετάσχουμε με τρόπο διαφορετικό από ό,τι σήμερα. Δεν θέλουμε διαρκώς να ζητούμε εμείς κονδύλια. Άρα τα ζητήματα αυτά έχουν όλα μεγάλη σημασία και πραγματικά ελπίζω να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ε, και να ενημερώσουμε σωστά τις κρατικές αρχές. Τέλος, να πω ότι ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ Υπουργείων είναι ένα σημαντικό θέμα. Αισθάνομαι πολλές φορές ότι το Υπουργείο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, το κατεξοχήν αρμόδιο για την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής από την Κροατία κάποιες φορές είναι απομονωμένο, χωρίς στήριξη από τα υπόλοιπα Υπουργεία. Αυτό το είδα να συμβαίνει και σε άλλα κράτη-μέλη. Μπορεί λοιπόν να προτείνουμε στη Λιθουανική Προεδρία όταν οργανώσει το άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο για την Περιφερειακή Πολιτική να μην προσκαλέσει μόνον Υπουργούς Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και τους Υπουργούς Οικονομικών. Διότι τουλάχιστον οι Υπουργοί αυτοί είναι από τους πρώτους που θα έπρεπε να συμμετέχουν επίσης στην όλη διαδικασία ελοποίησης της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ ιδιαίτερως. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ήταν ευτυχές που μπόρεσες να συμπληρώσεις αυτά που μας είπε ο κύριος Γκουλέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με συγχωρείτε, αλλά θα δώσω το, λόγο στον κύριο Κέλλη για ένα λεπτό, γιατί μόλις ήρθε και είναι καραδοκή για να πει κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχηθώ στην ε, Κροατία. Καλώς ήρθατε. Αλλά τι έχει να πει για την σύγκριση Κροατίας με τη δική μου τη χώρα, με παρόμοιο αριθμό πληθυσμού. Και όταν προσχωρήσαμε στην Ένωση πριν τόσα χρόνια, το ΑΕΠ μας ήταν περίπου αυτό της Κροατίας σήμερα. Με τις υποδομές μας όμως είχαμε μεγάλη βοήθεια από τα διευθυντικά ταμεία. Και άλλαξε πολύ η θέση μας όταν γίναμε κράτος μέλος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη σε αυτή τη στήριξη αφήσαμε πίσω μας την κέλτικη κληρονομιά μας. Βέβαια, τα... οι δυνατότητε τη Κροατία ω τώρα ήταν περιορισμένε, θα αυξηθούν πολύ με τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να γίνει συνετή αξιοποίηση των διευθυντικών κονδυλίων και των κονδυλίων συνοχή και πιστεύω ότι η Κροατία θα ε, προχωρήσει γρήγορα. Ελπίζω λοιπόν να είναι ένα από τα πληρέστερα, τα πλέον ενεργά και τα πιο επιτυχημένα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Ε, υπάρχουν τόσες αρνητικές στάσεις προς την Ευρώπη αυτή τη στιγμή που είναι θετικό να ε, προσχωρεί η Κροατία, η Λιθουανία να αναλαμβάνει την Προεδρία και η Λετωνία να, περνάει, να μπαίνει στην Ευρωζώνη. Είναι νομίζω μια ευτυχή στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένω να έχουμε μια καλή συνεργασία. Ε, πρόεδρος, ευχαριστώ Σον. Αλλά νομίζω, δεν θέλω χωρί να σα στενοχωρήσω, η δική του η ακτογραμμή είναι πιο ωραία και από τη δική σα. Αξίζει να την επισκεφθείς. Να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Γκουλέ και την Ιβάνα Μαλέτιτ. Είσαστε από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, σωστά, δεν είστε μαζί μας, αλλά ήταν καλό που ήρθατε. Περνάμε στο σημείο 19, τροποποίηση του κανονισμού για το άνοιγμα της αγοράς των χώρων επιβατικών συνδυοδομικών μεταφορών. Ρόζα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για τον κανονισμό που επέβαλε η Επιτροπή, μια τροποποίηση δηλαδή για τις εθνικές αρχές επιβατικών μεταφορών μέσω σιδηροδρόμων. Η πολιτική μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως γνωρίζετε, επικεντρώνεται στο να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός και να υπάρχει μια ισορροπία στις οικονομικές δραστηριότητες. Ο κανονισμός λοιπόν διευκρινίζει τις υποχρεώσεις των αρμόδιων δημόσιων αρχών και διευκρινίζει διάφορες πτυχές. Για παράδειγμα, προτείνει μέτρα για μεγαλύτερη διαφάνεια στην σχέση του ορισμού των υποχρώσεων των δημόσιων υπηρεσιών, γιατί όπως γνωρίζετε, όταν μία διαδρομή δεν γίνεται κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις, τότε οι κυβερνήσεις συζητούν για τα, τις διαδρομές αυτές που είναι κοινοφελούς ενδιαφέροντος να τα αναλάβουν οι πάροχοι ακόμα και αν δεν αποδίδουν. Έπειτα υπάρχουν και ποσοτικοί περιορισμοί για τις απευθείας αναθέσεις από... Δεν μπορεί να υπάρχει μετά από κάποιο διάστημα κανένας, καμία διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμβασης. Συμφωνούμε λοιπόν απόλυτα και νομίζω ότι οι γενικές αρχές της πρότασης είναι καλές. Με τις τροπολογίες μας προσπαθούμε να διευκρινίσουμε κάποια θέματα, είτε γλωσσικά είτε άλλα. Υπάρχουν κάποιες ασάφειες. Τι είναι δηλαδή ένας αστικός χώρος. Προσπαθούμε να πετύχουμε μια διευκρίνηση, έναν ορισμό ή τέλος πάντων ορισμός να είναι όπως ήταν και πριν ή ορισμός της αρμόδιας τοπικής αρχής, αρμόδια για τον κανονισμό, γιατί με τον νέο ε, ορισμό προκύπτει κάποια σύγχυση. Διευκρινίζουμε λοιπόν κάποιους όρους και ζητάμε κάποιες γλωσσικές τροποποίησεις. Πάντως, με δύο λόγια, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι θετική. Διατηρούνται οι περισσότεροι ορισμοί που υπήρχαν ήδη γιατί πιστεύουμε ότι είναι πιο ξεκάθαρη. Όπου υπάρχει ασάφεια ζητάμε διαγραφή των νέων όρων. Κατά τα άλλα, συμφωνούμε απόλυτα με την πρόταση. Να ξέρετε ότι η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος ενός γενικότερου πλαισίου που είναι το τέταρτο πακέτο σιδηροδρόμων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω εδώ σκιώδης αν δεν υπάρχει κανείς εδώ να αντικαταστήσει τους ε, Σκιώδης, περνάμε στους συναδέλφους. Ο κύριος Σόκη Βλάση. Α, είσαστε και Σκιώδης. Ωραία, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω τσεχικά, αν μου επιτρέπετε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προετοιμασία αυτής της πρότασης την οποία στηρίζουμε. Έχουμε όμως κάποιες επιφυλάξεις για αυτό το σιδηροδρομικό πακέτο και για το ότι πρέπει να καταλήξει σε άνοιγμα της αγοράς, σε περισσότερο ανταγωνισμό και χαμηλότερες τιμές για τους επιβάτες. Ε, αυτό και τους ε, πελάτες. Αυτό το στηρίζουμε βεβαίως, αλλά έχουμε κάποιες αμφιβολίες για τις συμβάσεις ε, μικρο όγκου γιατί υπάρχει δυνατότητα στις αρχές να μην προκυρήσουν διαγωνισμούς στην περίπτωση στην οποία το κόστος του διεξαγωγής του διαγωνισμού θα είναι μεγαλύτερο από το όφελος με διεξαγωγή του, Δηλαδή μιλάμε για μικροσυμβάσεις ε, κατ' ουσίαν. Όμως, αν γίνουν δεκτές τέτοιες προτάσεις, ανοίγει η πόρτα για κάποιες ε, πρακτικές ε, ε, σύμφωνα με τις οποίες θα δίνονται στις εθνικές εταιρείες πάρα πολλά μικρά συμβόλαια χωρίς διαγωνισμό. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να θέλει να μιλήσει. Μπορούμε να τελειώσουμε το ζήτημα. Εκτός εάν θέλει η Ρόζα να πει κάτι. Όχι. Θα μελετήσουμε αυτό που είπατε. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τίποτα άλλο. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Άρα το μόνο πρέπει να αποφασίσουμε είναι προθεσμία για τροπολογίες που θα είναι για Σεπτέμβριο. Γιατί η Επιτροπή Μεταφορών τέλει Νοεμβρίου έτσι κι αλλιώς δεν κρίνει την έκθεση αυτή. Οπότε 12 Σεπτεμβρίου ε, το μεσημέρι στις 12 είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Και περνάμε τώρα στο σημείο 20. Μαρή Τερές Σάντσε Σμιθ. Πρόκειται για την διαλειτουργικότητα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως είπε και η Ρόζα πριν, υπάρχει οδηγία για την διαλειτουργικότητα που αποτελεί μέρος του τετάρτου πακέτου σιδηροδρόμων. Όπως λέει και το όνομα της έκθεσης αυτής, είναι κάπως τεχνική, λίγο δύσκολο να σας την παρουσιάσω. Η Επιτροπή μας αποφάσισε να γνωμοδοτήσει. Και εγώ προσπάθησα να μελετήσω με λεπτομέρειε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δω τι βελτιώσει μπορούμε να επιφέρουμε. Παρά λοιπόν την τεχνική πτυχή, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαλειτουργικότητα στου σιδηροδρόμου είναι κάτι που συνδέεται με την εδαφική συνοχή, με την χωροταξία, και με τις διασυνοριακές ε, ανταλλαγές. Πράγμα που σημαίνει ότι η διαλειτουργικότητα πρέπει να επιτρέπει σε ένα βαγόνι να κυκλοφορεί σε οποιοδήποτε τμήμα του συνδρομικού δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς κανένα πρόβλημα. Και θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ξέρετε ότι εγώ προέρχομαι από την Νότια Γαλλία, ζω πολύ κοντά στα σύνορα με την Ισπανία. Εκεί έχουμε ένα τρένο υψηλής ταχύτητας από το Περπινιάν στην Βαρκελόνη, το οποίο δεν λειτουργεί αυτή την εποχή. Ενώ υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και δεν λειτουργεί λόγω έλλειψη διαλειτουργικότητα. Δεν μπορεί δηλαδή απευθεία το βαγόνι να πάει, ο σειρμό να πάει από το Περπινιάν στη Βαρκελόνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί με ενδιαφέρει όλου ιδιαίτερο αυτό το θέμα τη διαλειτουργικότητα. Δυστυχώ βρισκόμαστε ακόμα μακριά από μια κατάσταση όπου τα συστήματά μας θα ήταν απόλυτα αποτελεσματικά γιατί έτσι κι αλλιώς για ιστορικούς λόγους και επίτηδες τα σιδηροδρομικά δίκτυα φτιάχτηκαν διαφορετικά για να προστατεύσουν την εθνική επικράτεια για να αποφύγουν την εισβολή ξένων. Αυτό ήταν την εποχή του πολέμου. Σήμερα όμως δεν ισχύει πια. Έχουμε την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχουν πια τέτοιες απειλές. Καταργήσαμε τα σύνορα με τη συνθήκη, αποφασίσαμε ότι δεν υπάρχουν, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν. Ξεχάσαμε ότι τα σύνορα αυτά υπάρχουν στην καθημερινή ζωή των πολιτών και ότι οι υποδομές δεν είναι προσαρμοσμένες σε αυτό το άνοιγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν υπέβαλε το τέταρτο πακέτο σιδηροδρόμων τον Ιανουάριο με τη φιλοδοξία να ολοκληρώσει αυτόν τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο μειώνοντας συγχρόνως και το κόστος για τους ε, επιβάτες. Οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης αυτής για τα κράτη-μέλη, για τις περιφέρειες και για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τους επιβάτες με δύο λόγια, τους πολίτες, επιπτώσεις θα είναι τεράστιες. Η Επιτροπή μας λοιπόν αξιολογεί τις επιπτώσεις των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην συνοχή στην Ευρώπη και γι' αυτό και γνωμοδοτούμε. Στόχος λοιπόν της αναδιατύπωσης της οδηγίας αυτής για την διαλειτουργικότητα είναι να μειώσει τον κατακαιρματισμό και το κόστος για την κυκλοφορία των σειρμών και των βαγονιών. Και προκειμένου να έχουμε και τη μέγιστη ασφάλεια. Θα σας υπενθυμίσω λίγο τι γίνεται, πώς παίρνει άδεια λοιπόν ένα σειρμός ή ένα βαγόνι. Είναι περίπλοκο. Γιατί σήμερα η διαδικασία αυτή μπορεί να κρατήσει δύο χρόνια και να κοστίσει μέχρι 6 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 11.000 διαφορετικοί κανόνες ασφάλειας και κυκλοφορίας στην Ευρώπη. Η υπηρεσία σιδηροδρόμων μπορεί μόνο ρυθμιστικά να λειτουργήσει. Δηλαδή ορίζει τους κανόνες για να μειωθούν όσο γίνεται διάφοροι εθνικοί κανόνες. Συνεπώς, η άδεια για την κυκλοφορία των σειρμών είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Υπάρχουν τεράστιες αποκλήσεις για τον τρόπο με τον οποίο ακολουθούν τη διαδικασία διοδότησης οι εθνικές αρχές και επιστοποίησης. Σα είπα ότι μπορεί να κρατάει δύο χρόνια και να κοστίζει μέχρι 6 εκατομμύρια ευρώ μια τέτοια διαδότηση. Από τα νούμερα που έχουμε φαίνεται ότι η διαφορά είναι μέχρι 10% από χώρα σε χώρα. Όταν χρησιμοποιούνται σε τρει χώρε οι σειρμοί, μέχρι 30% μπορεί να φτάσει η διαφορά αυτή. Ορισμένε εθνικέ αρχέ αποφελούνται εξάλλου για να επιβάλλουν προστατευτισμό, ζητώντα όλο και περισσότερα δικαιολογητικά και καθυστερούν όλο και περισσότερο τι αδειοδοτήσει. Θέλουν να ξαναγίνουν δοκιμές οι οποίες έχουν ήδη γίνει όμως στο παρελθόν. Οι καινοτομίε λοιπόν τη ανδιατύπωση αυτή έχουν ω εξή. Η πρόταση τη Επιτροπής για ορισμένε χώρε είναι επαναστατική, γιατί καταργεί την εθνική αδειοδότηση και διατηρεί μόνο την άδεια για την κυκλοφορία. Και η μισορδομική υπηρεσία έχει την ευθύνη της κυκλοφορίας των σειρμών. Άλλη καινοτομία είναι ότι η Επιτροπή θέλει λειτουργική ευθύνη να αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός επιπλέον από το ρυθμιστικό του. Είναι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός που θα δίνει τις άδειε για την πρόσβαση στην αγορά αφού προηγουμένως πιστοποιήσει ότι το υλικό είναι σύμφωνο με τις διατάξεις και η πιστοποίηση αυτή θα ισχύσει ολόκληρη την Ευρώπη. Τεράστια πρόοδος. Οι εθνικές αρχές ασφάλειας, συνεπώς, δεν έχουν πια ευθύνη όσον αφορά την άδεια για τους σειρμούς. Αυτές είναι οι προτάσεις τροποποίησης που σας προτείνω. Εννοείται ότι με ενθουσιασμό υποδεχόμαστε τις προτάσεις της, Επιτροπής που, Επιτροπής που οδηγεί σε μια πραγματική απλοποίηση, την οποία και εμείς επιθυμούμε για να έχουμε έναν πραγματικά ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών όσον αφορά τις διαδικασίες του ετούντες και έτσι έχουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσέγγιση για την πιστοποίηση των σειρμών. Όμως ήθελα να τροποποιηθεί η διαδικασία για την πρόσβαση στην αγορά, γιατί νομίζω ότι εδώ επιλογεύουν κάποιοι κίνδυνοι. Οι περισσότερες τροπολογίες έχουν να κάνουν με το άρθρο 20 του σχεδίου οδηγίας, που είναι και το πιο σημαντικό. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποτιμάει μερικά πράγματα. Πρώτον, τη δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού να αντικαταστήσει 27 εθνικές αρχές ασφάλειας. Την ικανότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού να γνωρίζει όλους τους κανόνες που ήδη υπάρχουν. Σας είπα, 11.000 υπάρχουν. Και αμφισβητεί επίση και τη δυνατότητα του οργανισμού να προβαίνει σε πραγματικού ελέγχου. Επιπλέον, στην πρόταση τη Επιτροπή, το κόστο και η ευθύνη ε, είναι ευθύνη μόνο των συνδρομικών επιχειρήσεων. Ενώ εγώ πιστεύω ότι το κόστος αυτό θα είναι πολύ μεγάλο και θα αποθαρρύνει αυτούς που θέλουν να έχουν πρόσβαση στην αγορά. Ο γαλλικός οργανισμός ή ο γερμανικός οργανισμός σιδηροδρόμων ή άλλοι μικροί που θέλουν να επαληθεύσουν κατά πόσο το τρένο μπορεί να ενταχθεί στο δίκτυο. Ενώ η ευθύνη αυτή, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι ευθύνη του κατασκευαστή. Όσον αφορά τώρα την αρχιτεκτονική. Στις 10 Ιουνίου βρέθηκε κάποιο σεβασμό στο Συμβούλιο για ισορροπία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Διατησία και την Εθνική Πραγματογνωμοσύνη. Εγώ θέλω να επανέλθω στις ιδέες αυτές, γιατί όταν το Συμβούλιο κάνει κάτι καλό που δεν το κάνει πάντα, πρέπει να το λέμε και να δείχνουμε ότι συμφωνούμε. Συνεπώς, με τη νέα αυτή αρχιτεκτονική, ο οργανισμός αποτελεί μόνο απευθυντική θηρίδα για κάθε έγκριση χρήσης οχήματος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να αποφύγουμε κάθε διάκριση που δεν δικαιολογείται με τίποτα, ότι η ΕΤΟΝ οφείλει να διευκρινίσει κατά την αίτησή του τη ζώνη χρήσης του οχήματος. Ο οργανισμός ε, επίσης, ο ευρωπαϊκός, διεξάγει τον έλεγχο για τους ειδικού, μάλλον αναθέτει τους ειδικού ελέγχους στην αρμόδια εθνική αρχή. Η εγκύτητα πιστεύω ότι αποτελεί εγγύηση και για την απλοποίηση. Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους ένα μήνα για να ζητήσουν τα πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία και έχουν τέσσερις μήνες το αργότερο για να αξιολογήσουν και να εξετάσουν το φάκελο. Ο οργανισμός λαμβάνει στη συνέχεια την απόφασή του ανάλογα με τις γνώμες των εθνικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο φορέας προσφυγών είναι αρμόδιο για να διευθετήσει τις διαφορές μεταξύ του οργανισμού και των εθνικών αρχών. Επίσης, προτείνω ένα εθνικό μητρό. Συγγνώμη, αντί για τα 27 εθνικά μητρό, ένα ευρωπαϊκό μητρό οχημάτων. Χάρη απλοποίησης. Μόνο οι αλλαγέ που χαρακτηρίζονται μείζονες στα οχήματα επιβάλλουν νέα έγκριση. Η ανάλυση του κόστους και ωφέλειας μιας νέας τεχνικής απλοποίησης θα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά. Τα ανταλλακτικά τώρα των οχημάτων πρέπει επίση να αποτελέσουν αντικείμενο εναρμόνιση για να διοχετευθούν στην ευρωπαϊκή αγορά πιο εύκολα. Τέλο, ο οργανισμός οφείλει να διατηρήσει τον έλεγχο τη έγκριση των συστημάτων ERTMS με σκοπό την εξασφάλιση του συντονισμού τη εφαρμογή του συστήματο αυτού σε όλη την Ευρώπη. Τέλο, μια σημαντική καινοτομία αποτελεί δυνατότητα επέκταση τη ζώνη χρήση έως τον πλησιέστερο συνδρομικό σταθμό, χωρίς να εφίσταται η ανάγκη νέας διαδικασίας, εφόσον βέβαια τα συνδρομικά συστήματα είναι παρόμοια. Έτσι τα τρένα μπορούν να κυκλοφορούν και διασυνοριακά. Θέλω επίση να αφαιρθώ και στη μεταβατική περίοδο. Λαμβάνοντα υπόψη το μέγεθο των εργασιών προσαρμογή που πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και του Εθνικού, προτείνεται η παράταση τη περίοδου μεταφορά σε τρία έτη αντί για δύο. Ωστόσο, μετά την πάροδο δύο ετών, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει αιτήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τον οργανισμό, ώστε να ανταποκριθεί στι νέε του αρμοδιότητε. Συγγνώμη αν μακρηγόρησα, αλλά το θέμα είναι πολύ τεχνικό και ήθελα να σα έχω εξηγήσει τι τροπολογίε μου. Επίση, θέλω να σα πω ότι οι αυτοί κανόνε έχουν τεράστια σημασία για την εδαφική συνοχή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα μέσα της δεκαετίας 90. Το γεγονός ότι δεν έχει επενδύσει σε κάποιους τομείς η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση το 10 καταρχήν, δημιούργησε μια φθορά. Μια φθορά και του τροχαίου υλικού και των υποδομών με αποτέλεσμα οι σιδηρόδρομοι να έχουν γίνει λιγότερο ελκυστικοί. Η διαλειτουργικότητα όμως τώρα θα επιτρέψει να βγουν από την απομόνωση κάποιες ευρωπαϊκές περιφέρειες, να μειωθεί το κόστο για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, να επιταχυνθούν οι ανταλλαγές και να γίνουν πιο ελκυστικές σε διάφορες περιφέρειες στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε Μαρή Τερέζ. Δεν πρόσεξα ότι θέλω το λόγο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε η κυρία Στάρα θα λάβει το λόγο για να συμπληρώσει για το προηγούμενο σημείο μόλι ολοκληρώσουμε αυτό. Ο κύριο Βλάσακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, να ευχαριστήσω την κυρία Σάντε Σμιτ για την διεξοδική προετοιμασία της πρότασης και για την παρουσίαση που μας έκανε. Ήδη κάποιες απαντήσεις στις απορίες που ενδεχομένως να είχα, ε, ήδη έχω λάβει πολλές απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. η έγκριση για την κυκλοφορία των ε, οχημάτων αυτή τη στιγμή δίνονται από τους εθνικούς φορείς. Υπάρχουν ε, σοβαρές διαφορές μεταξύ των διαφορών απαιτήσεων ή των αιτήσεων πρέπει να υποβάλλονται κάθε φορά. Λόγω χάρη δοκιμές για τις τελευταίες ε, κινητήριες μηχανές που κατασκεύασε η Σκόντα. Τις μηχανές έλξης. Το 2012 ήταν ε, διαφορετικά τα πράγματα στη Γερμανία και με συγκεκριμένες απαιτήσεις. Θα έπρεπε να νομιμορφεί κανόνες παντού. Και το ερώτημά μου προς την κυρία Σάντσι Σμιτ είναι πότε θα μπορεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός να καλύπτει όλα αυτά τα ζητήματα. Διότι θα πρέπει να υπάρχει πλέον διασυνοριακή λήψη αποφάσεων από τις 27 αρχές ταυτόχρονα. Και έπειτα για το κόστο. Αυτή η ευρωπαϊκή αδειοδότηση πόσο θα κοστίζει. Εάν είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, ίσω να μην υπάρχουν αρκετέ αιτήσει, αρκετό ενδιαφέρον και για τη ζώνη χρήσης των οχημάτων. Ίσως αυτό θα πρέπει να το αποφασίσουμε σε διμερές επίπεδο. Σε μια πρώτη φάση αυτό θα ήταν λιγότερο δαπανηρό ενδεχομένως. Και όπως σωστά είπε η συγγήτρια, θα υπάρχουν και χρονικά περιθώρια. Ένας μήνας για την ε, εξέταση της αίτησης που έχει υποβληθεί και δύο μήνες για την αδειοδότηση, για τη χορήγηση της άδειας εάν η αίτηση οδεύει στη σωστή κατεύθυνση. Θα είναι μια περίπλοκη διαδικασία παρόλα αυτά. Οφείλουμε να γνωρίσουμε. Γι' αυτό καλό είναι η μεταβατική περίοδο να γίνει από δύο χρόνια, τρία. Αλλά ελπίζω όλα τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν σε αυτή τη συμφωνία και σε αυτό το σύστημα. Ιδάλω δεν θα έχει νόημα. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τη συνάδελφο για όλε τι λεπτομέρειε και τα ενδιαφέροντα στοιχεία που συμπεριέλαβε σε, αυτό, σε αυτή την πρόταση. Είστε κι εσείς κοιόδης εισηγητής, σωστά. Oui. Ναι. ναι, είμαι σκιώδης εισηγητής για το τέταρτο πακέτο για το τμήμα της ε, διακυβέρνησης. Δηλαδή θέλετε το λόγο τώρα. Ε, θα μιλήσω όταν μιλήσουμε για την διακυβέρνηση. Ναι. Τη διαλειτουργικότητα εννοείται με το κουβερνάω στα γαλλικά. Γιατί είναι τρία τα στοιχεία του ίδιου πακέτου. Ναι. ναι, και για τη διαλειτουργικότητα θέλω να μιλήσω. Για την έκθεση λοιπόν αυτή ως έχει στις αιτιολογικές σκέψεις βρήκα ότι υπήρχε έντονη τάση να γίνεται λόγος για την απελευθέρωση και την ανταγωνισμό, την ανταγωνιστικότητα μάλλον. Σε συγκεκριμένες όμως τροπολογίες, όπως έχουν υποβληθεί, δεν αντιλήφθηκα να γίνεται το ίδιο. Για την ώρα λοιπόν δεν έχω δει συγκεκριμένε παρατηρήσεις για τις τροπολογίες πέραν αυτής και θα φροντίσω να υποβάλω εκεί που χρειάζεται τροπολογίες, πάντως πέραν της γενική παρουσίαση. επί της οποίας έχω κάποιες ε, διαφωνίες ε, ε, επί έχω κάποιε διαφωνίε, θα, θα φροντίσω να υποβάλω τι κατάλληλε τροπολογίε για να συμπληρώσω τα κενά. Ε, ωραία, να ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον κύριο Πράουτ. Η κυρία Πράουτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Σάντζε Σμιτ, για την έκθεσή της, για τη διαλειτουργικότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι διεξοδική η έκθεση έτσι όπως την έχει ετοιμάσει ως προς τις τροπολογίες μάλιστα που έχει υποβάλει και οι τροπολογίες που αφορούν το ενιαίο Ευρωπαϊκό Μητρό για τα οχήματα. Εδώ συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι αυτό θα συνέβαλε στη δημιουργία ενός ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου για την Ευρώπη. Όμως μπορεί να υπάρξουν συνέπειες στους πόρους μας. Αυτό θα πρέπει να το πελετήσουμε, λοιπόν προηγουμένως για την μετάβαση σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα σήμανσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων είναι εκείνος που θα χορηγεί και τις άδειες για τη θέση σε λειτουργία των ε, διαφόρων ε, σιδηροδρομικών τροχιών και των συστηματών e ERTMS. Θα προτιμούσαμε λοιπόν η συγγήτρια να έχει μεγαλύτερες και η Επιτροπή σας να δείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία στο σημείο αυτό και να δώσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μεταβατική περίοδο και την ε, υλοποίηση της νέας διαδικασίας Ο ERA ήδη ετοιμάζεται για αυτές τις νέες ε, διαδικασίες ως προς τους πόρους εξετάζει πώς θα αρχίσουν ε, εκ των προτέρων να δοκιμάζονται και να υλοποιούνται. Θα θέλαμε λοιπόν επαρκή πρικοδότηση και συμφωνούμε ότι καλό θα ήταν να παραταθεί η μεταβατική περίοδος από τη διετία σε τριετία. Οπότε δεν συμφωνούμε με την τροπολογία της εισηγήτριας να γίνει η διετία τριετία. Θα θέλαμε να γίνουν όλα αυτά πιο σύντομα. Ως προς τις προθεσμίες φαίνεται να υπάρχει μια υποπροϋποθέσεις ε, μεταφορά. Κάτι όμως που θα δημιουργήσει κενό νομικό, αβεβαιότητα. Και δεν συνάδει με το γενικό μας στόχο να έχουμε ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα για τον τομέα των σιδηροδρόμων. Για τις υπόλοιπες τροπολογίες κάποιες είναι τεχνικής φύσης και θα πρέπει να μελετηθούν ε, αναλυτικά αλλά θέλουμε να υπάρχει συνεκτικότητα στο κείμενο. Λόγω χάρη η τροπολογία για τα ανταλλακτικά ή την υποχρέωση στα ETSI να εντοπίζονται τα ανταλλακτικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπέρ έτσι κι αλλιώς αυτής της προσέγγισης της τεχνικής προδιαγραφής διαλειτουργικότητας, οπότε αυτό θα πρέπει να το μελετήσουμε ίσως με ιδιαίτερη νομοθετική προσέγγιση. Προφανώς είναι αυτονόητο ότι όλες οι τροπολογίες που αφορούν την υλοποίηση με κατεξουσιοδότηση πράξης, εκεί υπάρχει τόσο άλλο γενική επιφύλαξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως κατά τα άλλα καλωσορίζουμε την πρόταση της εισηγήτρας ως έχει. Ευχαριστούμε. Μαρή Τερέζ, θέλεις να κλείσεις τη συζήτηση με κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνούμε νομίζω όλοι για την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τον κατακαιρματισμό του συνδρομικού συστήματος των κατομελών. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, το ανέφερε ο κύριος Βλάσοκ για τη χώρα του. Ε, ερωτήσεις, όχι εμφιβολίες, ερωτήσεις έχουμε για την ικανότητα του οργανισμού να αναλάβει όλες του τις ευθύνες, τόσο τεχνικές ευθύνες αμέσως. Αυτό με οδήγησε να ζητήσω παράταση της μεταπατικής περίοδου. Βέβαια, το, αυτό μπορούμε να το διαπραγματευτούμε. Θα δούμε την επιχειρηματολογία των μεν και των δε. Πάντως εδώ στο Κοινοβούλιο γνωρίζουμε την πραγματικότητα, πώ είναι τα πράγματα στην πράξη. Όπως είπε ο κ. Βλάσακ, θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να πάρουν μέρο σε αυτή την προσπάθεια να παίξουν το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι σήμερα οι κανόνε κάποιε φορέ είναι εργαλείο ή μέσο που επιτρέπουν και κάποιε τάσει προστατευτισμού να εκδηλώνονται. Εδώ έχουμε μια τεράστια πρόκληση όμω για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργηθεί ένα πραγματικό ε, Ευρωπαϊκό χώρο των συνδυοδρομικών μεταφορών. Σα ευχαριστώ πάντω που δεχτήκατε ευνοϊκά την πρότασή μου για το Ευρωπαϊκό Μητρό. Νομίζω ότι πραγματικά θα επιτρέψει να προχωρήσουμε προς τον ευρωπαϊκό χώρο που ανέφερα πριν και έπειτα με τους διαφόρους εταίρους και ενδιαφερομένους, τα κάτι μέλη δηλαδή, αλλά και τους ε, φορείς της εταιρείας υδροδρόμων θα δούμε πώς μπορεί να γίνει ακριβώς η υλοποίηση. Σαφώς ο Αντώνιο Ματσάδο, μεγάλος Ισπανός ποιητής, λέει ότι μαθαίνει κανείς να περπατάει περπατώντας. Άρα σε αυτή την ευρωπαϊκή μας προσπάθεια ε, αυτό το πνεύμα μας διαπνέει και νομίζω ότι αυτήν ε, την προσπάθεια κάνουμε όλοι. Αν μη τι άλλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην τωρινή περίοδο των τόσο μεγάλων αμφιβολιών και φόβων μπορεί σε τέτοια περιπτώσεις με το θέμα αυτό όπως Ευρωπαϊκός Χώρος των Συγκροδρόμων, να προσφέρει κάτι παραπάνω στην επιρροή της Ευρώπης. I would like to... Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω εδώ πέρα η προθεσμία για τις τροπολογίες να είναι η 12η Σεπτεμβρίου το μεσημέρι γιατί δεν βιαζόμαστε οπότε υπάρχει χρόνος για τροπολογίες και τώρα θα ήθελα να περάσουμε στο προηγούμενο θέμα της ε, ημερήσιας ε, διάταξης ε, να ζητήσω τον κύριο Λιεζουά να κάνει τις παρατηρήσεις του για την επόμενη Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την έκθεσή σας για αυτό το περίπλοκο θέμα που έχει να κάνει με την βελτίωση των υπηρεσιών και των σιδηροδρόμων. Πρόκειται για τις δημόσιες συμβάσεις βέβαια σχετικά με τους σιδηροδρόμους. Μας ενδιαφέρει επίσης όμως και η καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Αυτή λοιπόν είναι η στόχη των συμβάσεων ε, αυτών. Ο εισηγητής σας πολύ καλά εντοπίζει τα προβλήματα τα οποία τίθενται στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, ιδιαίτερα στην αγορά συμβάσεων δημοσίων υπηρεσιών. Ο προστατευτισμός των ιστορικών παρόχων δυσκολεύει, για να μην πω και εμποδίζει την πρόσβαση στην αγορά νέων παρόχων που θέλουν να παρέχουν νέες υπηρεσίες. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχουν πολλές λύσεις, χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και να γενικευτεί η διαδικασία διαγωνισμών. Θέλω όμως εδώ να εντοπίσω τρία σημεία σχετικά με τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυσκολεύεται να συμφωνήσει με τις τρολογίες της εισηγήτριας. Η πρώτη τροπολογία είναι η τροπολογία αριθμός 2, η οποία έχει να κάνει με τον ορισμό της αρμόδιας τοπικής αρχής. Και επιμένω στο τοπικής, το υπογραμμίζω. Ο ορισμός είναι πολύ σημαντικός και πρέπει κανείς να τον αντιληφθεί σε συνδυασμό με μια άλλη έννοια που είναι ο εσωτερικός πάροχος. Και τι είναι ο εσωτερικός πάροχος είναι αυτός ο οποίος ελέγχεται απευθείας από την αρμόδια αρχή. Ο κανονισμός λοιπόν προβλέπει τη δυνατότητα η αρμόδια τοπική αρχή να αναθέσει απευθείας, χωρίς δηλαδή διαγωνισμό, μια σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας σε έναν εσωτερικό πάροχο. Όταν πρόκειται για εξαίρεση, η εξαίρεση πρέπει να οριοθετείται πολύ συγκεκριμένα και γι' αυτό ε, με τον κανονισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αλλάζει, θέλει αυτή η άμεση, η απευθείας ε, ανάθεση να γίνεται μόνο στο τοπικό επίπεδο. Αν είχαμε τέτοιες αναθέσεις σε άλλο επίπεδο, πέραν του τοπικού, τότε θα είχαμε αρμόδιες αρχές οι οποίες θα ανέθεταν τέτοια συμβόλαια σε περιφερειακό επίπεδο ή ακόμη και σε επίπεδο πολλών περιφερειών για να μην πω και σε εθνικό επίπεδο. Κάτι το οποίο θα σήμαινε ότι τελικά δεν θα υπήρχε ανταγωνισμός γιατί τελικά λίγα συμβόλαια θα αναθέτονταν με διαγωνισμό. Δεύτερον, τροπολογία αριθμός 3 που έχει να κάνει με το πεδίο εφαρμογής και την έννοια του δικτύου. Εκπλήσεται η Επιτροπή που η συγγήτρια διαγράφει αυτή την τροποποίηση, αυτή την προσθήκη που θέλουμε εμείς στο νέο κανονισμό για τις υποχρεώσεις των ε, δημοσίων υπηρεσιών, γιατί η έννοια των δικτύων είναι πολύ θετική, κυρίως για την περιφερειακή πολιτική γιατί έτσι αναγνωρίζεται ότι μία σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας δεν είναι σύμβαση μόνο για μία γραμμή μεταφοράς, αλλά για ένα σύνολο γραμμών, για ένα δίκτυο που διαπέτει από συνοχή για να προσφέρονται ικανοποιητικέ υπηρεσίες μεταφορών σε ένα δίκτυο. Πρόκειται για την αναγνώριση της δυνατότητας διασταυρωμένης χρηματοδότησης μεταξύ δηλαδή γραμμών οι οποίες αποφέρουν κέρδη και αυτών που δεν αποφέρουν κέρδη. Άρα οικονομικά πιστεύουμε ότι έχει νόημα αυτή η προστίκη. Έπειτα, ο νέος ορισμός που προσθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο να περιορίσει το δίκτυο στο αναγκαίο και στο αναλογικό. Δηλαδή, ο στόχος μας είναι να υπάρχει καλή ισορροπία ανάμεσα στις συμβάσει δημοσίων υπηρεσιών εκεί που χρειάζεται και των εμπορικών υπηρεσιών εκεί όπου οι συμβάσει δημοσίων υπηρεσιών δεν ε, είναι απαραίτητε. Τρίτο σημείο. Πρόκειται για την τροπολογία εκείνη η οποία θέλει να αυξήσει τον τεμίνη μισόριο, τη δυνατότητα δηλαδή να ανατεθεί απευθεία σύμβαση, συμβάσεις δηλαδή που δεν έχουν μεγάλη σημασία για την αγορά. Η Επιτροπή προτείνει ως όριο τα 150.000 χιλιόμετρα ετησίως και η συγκήτρια προτείνει 1.500.000, κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν είναι λογικό. Ο κύριος Γκρός, εισηγητής της Επιτροπής Μεταφορών, είπε το de minimis που προτείνει η Επιτροπή να γίνει 500.000 χιλιόμετρα ετησίως, κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποδεχτεί συμβαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ και κατά τα άλλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στη διάθεση τη εισηγήτριας αλλά και στη διάθεση οποιοδήποτε μέλου τη Επιτροπή αυτή για να απαντήσει σε ερωτήσεις που ενδεχομένω έχετε. πρόεδρο. σε ευχαριστώ. Θέλεις να απαντήσεις μήπως? Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας εξηγήσω το γιατί των τροπολογιών μου αυτών. Πράγματι, η διαφάνεια είναι το βασικό, γι' αυτό και έχουμε την τροποποίηση του κανονισμού. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, όταν υποβάλαμε την τροπολογία 2 σε σχέση με τον ορισμό του τι είναι αρμόδια τοπική αρχή, είχαμε υπόψη μας ότι ο σημερινός ορισμός του κανονισμού ήταν ικανοποιητικός. Γιατί στο νέο κανονισμό προστίθεται ένας ε, όρος για την αστική, την ε, ε, περιοχή της Υπέθρου που θεωρήσαμε ότι προκαλεί σύγχυση. Εμείς θεωρήσαμε ότι ο προηγούμενος ορισμός ήταν ικανοποιητικός. Για την τροπολογία 3 τώρα, σχετικά με τις ε, επιπτώσεις του δικτύου, οι δημόσιες υπηρεσίες πράγματι πρέπει να είναι συμβατές και να διατηρούν ισορροπία με τα εμπορικά δίκτυα. Γι' αυτό και ακριβώς όταν ο σημερινός ε, ορισμός είναι σαφής, μιλάει για τις δημόσιες αρχές, δεν δημιούργησε σύγχυση όσα χρόνια εφαρμόστηκε. Γι' αυτό με αυτό το καινούριο που βάζει για το τι αποκλείεται από τις δημόσιες υπηρεσίες και μιλάει για τις επιπτώσεις επί των δικτύων των εθνικών ή μη εθνικών περιφερειακών τοπικών κτλ. Δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς εννοεί με τις επιπτώσεις επί του δικτύου θεωρούμε ότι δεν είναι σαφές. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουμε σε κάτι. Όσον αφορά τώρα την τροπολογία 6 που αναφέρει τον αριθμό των χιλιόμετρων, θα δούμε μέχρι το Σεπτέμβριο τι τροπολογίες θα έχουν υποβληθεί και θα καταλήξουμε τότε, γιατί άλλα λένε οι αλλά άλλος θα καταλήξουμε. Καλώς, περνάμε τώρα στο τελευταίο τμήμα του πακέτου αυτού, ο ο κύριος Τσίλερ. Πρόκειται για την... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα αναφερθώ και εγώ σε αυτό το οποίο μόλις είπαν η Ρόζα και η Μαρή Τερέζ ότι δηλαδή ακριβώς ε, στους σιδηροδρόμους ε, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ενότητα να αναφέρω δύο μικρές ιστορίες. Το 97-98 ε, ήταν στο γραφείο μου ο δήμαρχος του Πόσναν, ο κύριος Γκρομπέλνη ναι, και συζητούσαμε βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ενότητα μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου για το ότι χρειαζόταν τότε αμέσως τη διεύρυνση Ευρωπαϊκή Ένωση με Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία κτλ. αλλά απόδειξη για το ότι υπήρχε Ευρωπαϊκή Ενότητα και υπάρχει Ευρωπαϊκή Ενότητα. Μιλάμε για ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών και πρέπει να υπάρχουν τη δυνατότητα να κινηθούν βεβαίω. Η κινητικότητα είναι βασικό σημάδι της κοινωνίας μας και η πρότασή μου ήταν πω ε, ε, Ευρωπαϊκή Ενότητα θα ήταν να υπάρχει η δυνατότητα να κυκλοφορεί ξανά το λεγόμενο τρένο του θεάτρου μεταξύ Πόσναν και Βερολίνου. Έπαιρναν τότε το τρένο από το Πόσναν, έβλε, μετά 5 ώρα το απόγευμα, έβλεπαν την παράσταση στο Βερολίνο και μετά τα μεσάνυχτα πήγαιναν στο ε, Πόσναν και το άλλο πρωί στη δουλειά. Ίσως λίγο πιο ξενυχτισμένοι. Όταν λοιπόν ξαναλειτουργήσει αυτό το τρένο θα έχουμε ευρωπαϊκή ενότητα και βεβαίως απέχουμε πολύ από αυτό. Επόμενο παράδειγμα. θα επισκεφθεί η Επιτροπή Συγκοινωνιών την Δυτική Πολωνία για να δει τις ε, συνδέσεις ε, τις συγκοινωνιακές με τη Γερμανία. Θα ξεκινήσουμε από το Κατόβιτσε. που απέχει 600 χιλιόμετρα από το Βερολίνο και βεβαίως εγώ ήθελα να πάω με το τρένο. Αλλά πιο γρήγορα πάει κανείς στη Νέα Υόρκη ε, από το Βερολίνο παρά στο Κατοβίτσε. Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση. Είτε μέσω Στσέτιν είτε Βαρσοβίας πρέπει να πάει και να κάνει τουλάχιστον 9 ώρες ή πρέπει να αλλάξει 3-4 τρένα όλα αυτά είναι σκάνδαλο και δείχνει πως ακριβώς το μεταφορικό εκείνο μέσο το οποίο λέμε πως ε, πληρώνει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι φιλικό προς το περιβάλλον και τα απέχει ακόμα πολύ από το να είναι πραγματικά ευρωπαϊκό. Και έχουμε τώρα το τέταρτο συντηροδρομικό πακέτο, και πάλι συζητάμε το θέμα της ε, διαλειτουργικότητας όπως είπε η Μαρή Τερέζ επικρατεί προστατευτισμός ε, κάποια στιγμή πρέπει να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι και να πούμε πως ε, πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν τα τρένα χωρίς εθνικούς εγωισμούς κτλ. Εδώ όμως είναι το μεγάλο αλλά Όσον αφορά λοιπόν τα συνοριακά δρομολόγια συμφωνούμε, αλλά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Ε, νομίζω πως ειδικά σε αυτά τα δρομολόγια πρέπει να υπάρξει μια προσαρμογή σε απαιτήσει των καιρών, αλλά και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο έχουμε τοπικούς σιδηρόδρομους ε, που είναι, έχουν γραμμές ε, μικρού πλάτους ε, γιατί δεν είναι καν συνδεδεμένα στο εθνικό δίκτυο. Οπότε πρέπει να υπάρχει και χώρος για την επικουρικότητα και να μην ισοπεδώσουμε τα πάντα με έτσι έναν τρόπο ευρωπαϊκό. Εκεί όπου λειτουργούν τα πράγματα και υπάρχουν ειδικέ ε, τοπικές συνθήκες, ξέρουν οι άνθρωποι καλύτερα τι χρειάζονται νομίζω από μας. Σε ανάλογη κατεύθυνση λοιπόν πηγαίνουν ε, και οι τροπολογίες μου και παρακαλώ τους συναδέλφους να δώσουν λίγο βάρος. Ελπίζω να έχουμε λοιπόν τροπολογίες, αναμένω τη συζήτηση με τους κοιόδης και μετά θα προσπαθήσουμε μαζί με τους συναδελφούς να τις ε, περάσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζαν Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να χαιρετήσω το έργο του εισηγητή που πραγματικά εστιάζει στην καλύτερη, στη μεγαλύτερη συμμετοχή των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Επειδή είμαι σκέφτης εισηγητής το θέμα, για το θέμα αυτό στην Επιτροπή Μεταφορών για τη διαχείριση των συνδρομικών υποδομών θα πρέπει να ε, έχουμε μια συνολική προσέγγιση με σεβασμό το αρχής της επικουρικότητας και των γενικών κανόνων της. Δηλαδή κάθε σύστημα να μπορεί να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του αντί να επιβάλλεται ένα ενιαίο μοντέλο. Είναι κάτι που θέλω να πω εδώ και το οποίο το βρίσκω θεμελιώδου σημασία. Ναι στο διαχωρισμό των ε, βασικών λειτουργιών, διότι αυτές ακριβώς μπορεί να είναι πηγή διακρίσεων εάν δεν γίνει σωστός διαχωρισμός και δεν θα υπάρχει και απόλυτη διαφάνεια των οικονομικών ροών. Βεβαίω, θα πρέπει τα, τα κέρδη από τη χρήση των υποδομών να πηγαίνουν προ το φορέα ώστε να μπορεί να χρηματοδοτεί τι δραστηριότητε για την τόνιση τη ανταγωνιστικότητα. Και ναι στι δημόσιε επενδύσει, την στήριξη των υποδομών για την επιδίωξη στρατηγικών στόχων. Με να ρυθμιστεί που ε, θα έχει ιδιαίτερε αρμοδιότητε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα μπορεί να διαχειριστεί τι διαφορέ ε, για τι διασυνοριακέ μεταφορέ. Όμω, έχοντα διαβάσει την πρόταση, δεν νομίζω ότι ο κάθετο διαχωρισμό είναι κάτι που το προτείνει ακριβώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι η καλύτερη ε, οδό για να υπάρξει μεγαλύτερη στροφή προς, τον, ε, προς τους σιδηροδρόμους μεν, από την άλλη όμως ο εισηγητής ζητά μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες λειτουργούν σε μικρότερα δίκτυα. Το σημειώνω αυτό. Επίση, καλό είναι να μεταφέρονται τα κέρδη από τη χρήση των αποδομών προ του φορεί. Αυτό το ε, Λέει ξεκάθαρη οδηγία και εκεί συμμερίζομαι το στόχο αυτό για τη συμπερίληψη των ευθυνών των εκπροσώπων των αρχών τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι με τα συμβούλια παρακολούθηση και στην όλη διαδικασία λήψη αποφάσεων είναι καλό να γίνει αυτή η επιλογή. Όμω θα πρέπει να βελτιώσουμε την πρόταση ω προ αυτό, ιδίω στην τροπολογία 7. Αυτό θα θέλω να το συζητήσουμε βάσει τη αρχή ότι η απόφαση διαχωρισμού θα πρέπει να είναι λιγότερο αυστηρή και θα πρέπει να είμαστε κι εμεί συνεπέστεροι ω προ τη διαδικασία που έχουμε προκρίνει. Δηλαδή, να μην ε, ε, παραμείνουμε στα κατάλληλα ενό συστήματο που ακόμη δεν είναι διαχωρισμένο σωστά. Θα πρέπει οι πολιτικοί θύνονται σε τοπικό επίπεδο να έχουν και το δικαίωμα να επηρεάσουν τη διοργάνωση του τοπικού συνδυοδρομικού δικτύου, διότι αυτή είναι υπεύθυνη από πολιτική πλευρά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη ευελιξία ακριβώ για να ανταποκρίνεται το συνδυοδρομικό δίκτυο στι ιδιαίτερε ανάγκε τι τοπικέ. Και για τι διαπεριφερειακέ μεταφορέ, τι διασυνοριακέ, θα πρέπει προτεραιότητα να δοθεί ακριβώ αυτή τη διασύνδεση, ώστε η όλη μεταρρύθμιση να είναι αποτελεσματική σε ευρωπαϊκό επίπεδο για του Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ότζι. Eh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή. Οπωσδήποτε κάποια πράγματα πρέπει να τα εξηγήσουμε καλύτερα. Εγώ την χάνει να είμαι σκιώδης ηγητής ε, για την τροποποίηση αυτής της οδηγίας. Οπότε το έχω μελετήσει το θέμα εδώ και καιρό. Βεβαίω, πρώτος στόχος πρέπει να είναι η απελευθέρωση. Γιατί θέλουμε οικονομικές ε, μεταφορές που θα είναι πραγματική εναλλακτική στις οδικές. Πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχει η διακριτική μεταχείριση εις βάρος ε, των μικρών ε, εταιριών και βεβαίως ε, καμία διακριτική μεταχείριση κανένας κράτους μέλους. Η πρόταση της Κομισιόν είναι να υπάρξει μια δομή holding μιας εταιρείας δηλαδή συμμετοχών για τις χώρες εκείνες που θα έχουν ήδη μια τέτοια δομή όταν τεθεί η ισχύ οδηγία. Αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή αν ε, μπορεί να το κάνουν αυτό κάποιες χώρες πρέπει να μπορούν να το κάνουν ε, όλες. Μετά για τις μικρές εταιρείες με λιγότερους από 50 υπαλλήλους σε ιστορικές γραμμές, τοπικές γραμμές, ε, με γραμμές ε, μικρού πλάτους κτλ. Δεν έχω καμία επιφύλαξη, αλλά και πάλι το ίδιο ε, με ό,τι και πριν. Δηλαδή, η εξαίρεση να δοθεί σε όσους ε, εκπληρώνουν αυτές τις συνθήκες. Εδώ πέρα λέτε μέχρι να τεθεί νησική οδηγία. Όχι, και μετά. Και στο μέλλον. γιατί σε πολλές περιπτώσεις είναι οι τοπικές αρχές οι οποίες είναι ε, αυτές που διαχειρίζονται τις γράμμες αυτές. Αυτά όσον αφορά τις επιφυλάξεις μου, ελπίζω να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ και η Κομισιόν, η κυρία Κράουτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και την Επιτροπή σας για το ενδιαφέρον που δείχνετε και βεβαίως αυτό δείχνει τι σημασία έχει ο σιδηρόδρομος για την εδαφική συνοχή. Έχουμε ένα φιλόδοξο εδώ πέρα πακέτο με στόχο την ολοκλήρωση της του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου με καλύτερη ποιότητα και περισσότερες επιλογές. Το τρέχον ε, νομικό πλαίσιο δεν επαρκεί για αυτές τις προκλήσεις. Η διαλειτουργικότητα όπως ακούσαμε δεν είναι πλήρης. Τεχνικοί κανόνες και κανόνες ασφαλείας είναι πολύπλοκοι και κοστίζουν πολύ οι διαδικασίες. Κατόπιν ο κλάδος ακόμα δεν επιτρέπει την βέλτιστη διαχείριση των υποδομών. Και τέλος μόνο οι εμπορευματικές μεταφορές και οι διεθνείς επιβατικές μεταφορές είναι ανοιχτές στον ανταγωνισμό. Οπότε μεγάλο κομμάτι των εσωτερικών αγορών είναι εθνικό μονοπόλιο. Η Κομισιόν έχει εξετάσει προσεκτικά την κατάσταση και τις διάφορες αγορές και έχει αξιολογήσει τον αντίκτυπο των διαφόρων επιλογών. Θα θέλαμε λοιπόν να καλωσορίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης που σε γενικές γραμμές στηρίζει το στόχο της Κομισιόν για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υποδομών. Σαφώς ο διαχωρισμός είναι απλούστερη και αποτελεσματικότερη λύση για να υπάρξει η συμμεταχείριση και πρόσβαση στη συνδρομική αγορά. Για να υπάρξει κάποια ευελιξία, παρόλα αυτά προβλέπουμε μια εναλλακτική επιλογή για τις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν τέτοιες δομές όταν θα τεθεί ενισχύ η συγκεκριμένη οδηγία. Βεβαίως η δεύτερη επιλογή είναι αποδεκτή για την Κομισιόν αλλά και για τα περισσότερα κράτη-μέλη εάν υπάρξουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας για να μην υπάρξει ακριβώς στρέβλωση του ανταγωνισμού. Καλώς ορίζουμε λοιπόν τις τροπολογίες του εισηγητή για την ενίσχυση των κανόνων δημοσιονομικής διαφάνειας ε, και οτιδήποτε ενισχύει την πρότασή μας. Θέλω όμως να πω πως έχουμε δύο σημαντικές επιφύλαξεις ή παρέκκληση που προβλέπεται για μικρές και καθετοποιημένες εταιρείες και για συγκεκριμένα επενδυτικά έργα πάει πάρα πολύ μακριά και τα κριτήρια δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τον αντίκτυπο στη λειτουργία της αγοράς κάποιες σχετικά μικρές υποδομές μπορεί να έχουν στρατηγική σημασία για τη λειτουργία της διαδρομικής αγοράς. Παραδείγματο χάρη είναι το τούνελ της μάχης. Μην ξεχνάμε ότι η Κομισιόν έχει κινήσει τη διαδικασία επί παραβάση. Γιατί πραγματικά είναι ε, στρατηγική σημασία για την ευρωπαϊκή σιδηροδρομική αγορά και υπάρχουν κάποια εμπόδια και θα πρέπει άρα παντού να υπάρχουν οι ίδιοι για να μην υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Για έργα υποδομής μικρής κλίμακας που δεν έχουν στρατηγική σημασία υπάρχει ήδη μία εξαίρεση στην ε, υφιστάμενη οδηγία την 2012-34 που υιοθέτησε πέρυσι το Κοινοβούλιο. Επίσης έχουμε προβλέψει μία διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης για να επιτρέψουμε στην Κομισιόν κατόπιν ετήματος κράτους μέλους ε, ή με δική της πρωτοβουλία να επαληθεύσει το εάν υπάρχουν ε, απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας σε καθετοποιημένες ζωμές. Προτείνει ο εισηγητής να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα περιορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης από πλευράς κρατών μελών και εδώ πραγματικά περιορίζεται το δικαίωμα που δίνει δυνατότητα να υπάρχουν ώρα ανταγωνισμού. Όσον αφορά τώρα την εμπλοκή των αρμοδίων τοπικών και εθνικών αρχών, η Κομισιόν ε, την στηρίζει καθώς είναι βεβαίως μεγάλοι πελάτες και χρήστες των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και ε, θα προωθήσουν οπωσδήποτε την καλύτερη ποιότητα παρόλα αυτά. Πρέπει να υπάρχει απαραίτητη ευελιξία και να μην είναι πολύ βαρκίνητες οι δομές. Ο συγητής επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλες φιλοδοξίες για τα εισιτηρία. Συμφωνεί επίσης ε, στους στόχους ε, και εμείς συμφωνούμε στους στόχους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, αλλά θα πρέπει να υπάρχει εμπορική ελευθερία καινοτομία των εταιριών. Και επίσης ίσως είναι πιο ρεαλιστικό να γίνει μια διάκριση μεταξύ ε, ολοκληρωμένης έκδοσης εισιτηρίων και ελεύθερης ε, έκδοσης εισιτηρίων. Τέλος, η τροπολογία υπαριθμών 10 που μιλάει για διαχειριστές ε, των υποδομών, η Κομισιόν δεν βλέπει κάποιο λόγο να καθυστερήσει η εισαγωγή του φορέα αυτού, καθώς μόλις όπως είπε ο εισηγητής τα προβλήματα υποδομών πύχη μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας ε, υπάρχουν γι' αυτό ακριβώς ε, και γι' αυτούς ακριβώς λόγους θέλουμε και εμείς να ε, δημιουργήσουμε αυτό το θεσμό Α, καλωσορίζουμε βεβαίως την φιλοδοξία του εισηγητή. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρος Γιώκημ. Θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο που είδε την έκθεση με τον καλό συνάδελφο Όλτριχ ε, για το επίμαχο ζήτημα. Νομίζω πως μπορούμε να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση για την παρατήρηση της Κομισιόν. Διαφωνώ, αλλά συμφωνώ με την αρχή Think Big, Act Local δηλαδή οι μεγάλες υποδομές που είναι στρατηγικές για τη λειτουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου ε, θα πρέπει να υπάρχει για αυτές μια πανευρωπαϊκή ρύθμιση της πρόσβασης αλλά εκεί πραγματικά όπου μιλάμε για σιδηρόδρομους τελείως διαφορετικής ε, μορφής ε, και χαρακτήρα δεν νομίζω πως χρειάζεται να ασχολείται με αυτά η Ευρώπη επαρκή η εθνική και η περιφερειακή αρμοδιότητα. Αυτά τα οποία επικομισιόνται τα σημείωσα και θα αντιδράσω αναλόγως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Οπότε πρέπει να ορίσουμε μια προθεσμία για τροπολογίες. Προτείνω την ίδια 12 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η επόμενη συνεδρία είναι 23 και 24 Σεπτεμβρίου. Άρα λύεται η συνεδρίαση. Εύχομαι καλές διακοπές σε όσους έμειναν μέχρι τώρα. Και, όπως είπα, λύεται η συνεδρίαση. Γεια σας.